Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν εχθές ε, στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση. Πραγματικά σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, διότι εχθές ξέρω ότι είχαμε πολλές συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες συμμετέχετε και παρόλα αυτά είχαμε σημαντική εκπροσώπηση από αυτούς τους λίγους που είμαστε πάντα στην Επιτροπή Αλίας και η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όπως ε, συνήθως γίνεται με αυτά τα πράγματα, όταν έχουμε πολύ κόσμο και πρέπει ο καθένας να μας πει την άποψή του. Ε, χάρηκα πολύ που είχαμε εδώ μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και στο μέλλον θα δούμε κατά πόσον μπορούμε να συνεχίσουμε με το σύστημα αυτό και κατά πόσον μπορούμε να το πλαισιώσουμε με διαφορετικό τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό. Φαντάζομαι ότι όσοι έλειπαν εχθές ε, είχαν τους λόγους τους, αλλά ευχαριστώ και πάλι τους παρόντες εχθές ε, και για τη συνεργασία και για τη συνεισφορά τους. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη καταρχάς και να περάσουμε στο σημείο 4 που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 7ης και 8ης Απριλίου του 2010. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, μέχρι το πέρας της σημερινής συνεδρίασης ε, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Στις ανακοινώσεις της Προέδρου δεν έχω και τίποτα να σας ανακοινώσω, επομένως να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 6, ψηφοφορία για τη χρήση στην ιδετοκαλοέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. Εισηγητής ο κύριος Φερέιρα και να του δώσω το λόγο σε περίπτωση που θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ιδάλω μπορούμε να ψηφίσουμε απευθείας. Κύριε Φεραίρα θέλετε το λόγο ή να ψηφίσουμε. Δεν ε, ενδιαφέρεται να παρέμβει ο κύριος Φεραίρα, επομένως ψηφίζουμε. Να ψηφίσουμε την τροπολογία 3 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Αυτό είναι. Δεκαοχτώ όλοι υπέρ. Ή κάνω λάθος. Η τεχνολογία πάλι μας προδίδει. Ε, ε, λοιπόν, 18 ψηφίσαντε και οι 18 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. και οι 18 ψηφίσαντε είναι υπέρ, εγκρίνεται. Στη συνέχεια, προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Το κείμενο το έχετε στον κατάλογο ψηφοφοριών, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συνέχεια, τροπολογία 15 δεν ψηφίζεται γιατί είναι γλωσσικού περιεχομένου και ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβιβαστική τροπολογία στο άρθρο 1 σημείο 2α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 16, 17, 18, η 5 του εισηγητή απεσύρθη. Επομένως ψηφίζουμε την 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 6 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφόρια. Εγκρίνεται. Από την 7 Μέχρι την ε, τροπολογία 13 ψηφίζουμε μπλοκ. Αυτό είναι το θέμα της επιτροπολογίας, ε, σε περίπτωση που δεν είναι σαφές για κάποιον. Το θέμα της επιτροπολογίας ψηφίζεται από κοινού, από το 7 στο 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνονται ομόφωνα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τέλος τροπολογία 2. με την προφορική τροπολογία. Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και επομένως ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Φερέιρα. Έχετε καταφέρει να έχετε ομόφωνη έγκριση έκθεση εδώ στην Επιτροπή μας. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση του κυρίου Κούν για θέματα επιτροπολογίας. Έκθεση Κούν. Η πρόεδρο δεν έχει τον κατάλογο ψηφοφοριών. Bueno, eh, en cualquier caso. Se propone un, un, en bloque. Ah, se propone un, un, un voto en bloque. Ah, vale, vale, vale. Προτείνεται να ψηφίσουμε μπλοκ. Κύριε Κούν, θέλετε το λόγο πριν ε, ψηφίσουμε την έκθεσή σας ή μάλλον τη γνωμοδότησή σας. Δεν θα ήθελα να, γίνω, να μην είμαι δημοφιλή στου συναδέλφου. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει. Είναι πολύ δύσκολο το πεδίο εργασία. Οι νέε συνθήκε εργασία μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, όπου ε, ε, βάση της, όπου η ετρυπολογία μετατρέπεται σε ε, πράξεις κατ' εκπροσώπηση, um πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. πρόκειται για το ζήτημα εξέτασης των εκτελεστικών διατάξεων που θα θεσπίσει η Επιτροπή είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτής της ειδική επιτροπής όπου εμπειρογνώμονες των χωρών μελών παρίστανται εκ μέρους του Συμβουλίου καθώς και οι υπάλληλοι της Επιτροπής εμείς θα έπρεπε να έχουμε το καθεστώς του παρατηρητού στο μέλλον. Αυτό αναφέρεται στις τροπολογίες και έτσι μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις πληροφορίες και να παραμβαίνουμε εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Έτσι μπορούμε να κάνουμε σωστή χρήση των κοινοβουλευτικών μας δικαιωμάτων. Δέχεστε να ψηφίσουμε αν μπλοκ όλες τις τροπολογίες του κυρίου Κούν. Δεν ε, βλέπω καμία αντίρρηση. Ψηφίζουμε αν μπλοκ. Ε, κύριε Ρόντου. Παρακαλώ. Εμείς θέλουμε να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία. Ωραία, να ψηφίσουμε ξεχωριστά λοιπόν. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 11 ψήφους. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 15 ψήφου. Τροπολογία 11. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 14 ψήφους. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται με 14 ψήφους. Τροπολογία 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. εγκρίνεται με 13 ψήφους. Η τροπολογία 14 απεσύρθη. τροπολογία 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 11 ψήφους. Τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με 11 ψήφους. Τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 14 ψήφους. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 15 ψήφους. Άρχεται ψηφο... Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 15 ψήφους. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 11 ψήφους. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Κούν. Σήμερα δίνουμε συγχαρητήρια σε όλους. Όλα γίνονται εδώ ανέμακτα. Ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 8. Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Χιλή για τη διατήρηση των αποθεμάτων ψηφία στον Ανατολικό Ειρηνικό Κενό. Εισηγητή ο κύριο Γκάλαγκερ. Και σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε την παρουσίαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε αυτό το μνημόνιο συμφωνία. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Νικολόβα. Νικολόβα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρουσίασή μου Αναφερόμενοι σε αυτήν την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής και για το λόγο τον οποίο ήταν σημαντική, η όλη ιστορία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν ευρωπαϊκά σκάφη με ισπανική σημαία δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα λιμάνια της Χιλής και ειδικότερα ε, μιλάω για σκάφη του ε, νοτιοδυτικού ε, ειρηνικού και τότε ο κλάδος ε, της Ισπανικής Αλίας έκανε προσφυγή γιατί αποτελούσε εμπόδιο εμπορικό για, τους, για τα ισπανικά σκάφη και στη συνέχεια υπήρξε έρευνα με πόρισμα ότι όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο, δηλαδή η απαγόρευση, απαγόρευση εκφόρτωσης ξηφία στα ε, λιμάνια της ε, Χιλής ε, κρίθηκε απαράδεκτη στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ξεκινήσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία διαδικασία στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά της Χιλής για το θέμα αυτό και στη συνέχεια ως αντίπεινα η Χιλή προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κοινότητας τότε. Το 2001 υπήρξε πολιτική συμφωνία μεταξύ της ε, ε, του Υπουργού Αλίας της Χιλής ε, και του Επιτρόπου ε, Αλίας να ανασταλεί η διαδικασία που έχει αρχίσει στο πλαίσιο του Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας για να υπάρξουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ Χιλής και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αποτέλεσμα αυτής ε, της, ε, αυτού του διακανονισμού ήταν ε, η συμφωνία του 2001 που, που επέτρεπε περιορισμένη πρόσβαση κάποιων ευρωπαϊκών σκαφών στους λιμένες της Χιλής και προέβλεπε κάποια πολυμερή διαβούλευση όσον αφορά τα αποθέματα του ξηφία, όπως επίσης και διμερή επιστημονική και τεχνική επιτροπή. Όσον αφορά αυτήν την τελευταία επιτροπή ε, και την πολυμερή ε, συμφωνία, λειτουργήσαν καλά. Ήταν πολύ επικοδομητική η συνεργασία και οι συζητήσεις μεταξύ ε, των δύο ε, μερών. Αλλά όσον αφορά την πρόσβαση των ε, κοινοτικών σκαφών στους λιμένες της Χιλής, αυτό ήταν ένα δύσκολο ζήτημα και τελικά δεν εφαρμόστηκε η συμφωνία η σχετική μετά τα πνεύματα οξύνθηκαν μεταξύ Χιλής ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γι' αυτό έπρεπε να επεξεργαστούμε περισσότερο τη συμφωνία του 2001 και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο ώστε να μπορέσει τελικά αποτελεσματικά να ε, συνεισφέρει στην διαχείριση των αποθεμάτων του ξηφία όπως επίσης και τη δυνατότητα εκφόρτωσης ξηφία στους λιμένες της Χιλής. Τον Απρίλιο του 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ε, για την νέα ε, συμφωνία με την Χιλή όσον αφορά την διατήρηση των αποθεμάτων του Ξηφία και έχετε μπροστά σας ε, το, την έκβαση των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα σε διάφορα στάδια. Και η συμφωνία, όσα έχει αυτή τη στιγμή, βασίζεται σε ό,τι υπήρχε ήδη το 2001, στο βαθμό βέβαια στο οποίο ε, ήταν επιτυχή όσα αναφέρονταν στη συμφωνία αυτή. Είναι πολύ πιο λεπτομερής η διαδικασία για την πρόσβαση στους λιμένες της Χιλής. Ε, βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα ε, στα μέτρα που ενέκρινε προσφάτως ο ΦΑΟ. Θα ήθελα λοιπόν δύο ε, πτυχές ε, να αναφερθώ, κυρίως στο 4 και στο 5 του Μνημειονίου Κατανόησης υπάρχει αναφορά των ε, αρμοδιοτήτων της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής και σκοπός μας είναι να υπάρχει ένα επίπεδο επιστημόνων, ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και συζήτηση της κατάστασης των αποθεμάτων και το δεύτερο επίπεδο στο οποίο θα συνέρχεται η Επιτροπή είναι ε, οι διευθυντές ε, που θα αποφασίσουν επί τη βάση των συστάσεων ε, των εμπειρογνώμων των, επιστημόνων κατά πόσο πρέπει να υπάρξει απόφαση διατήρησης των αποθεμάτων. Προβλέπει λοιπόν πρόσβαση για τα ευρωπαϊκά σκάφη αλίευσης ξηφία στην Αρίκα, στην Τουφακάστα και στην Πούντα Ρένα, τρία λιμάνια της Χιλής, ε, στην, ε, στις ακτές της ε, Χιλής, βορείος, νοτίος και το τρίτο είναι κάπου στη μέση. Τα τρία αυτά λιμάνια θα είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση, εκφόρτωση, επιδιόρθωση, επισκευής σκαφών και σε μερικές περιπτώσεις βέβαια ανωτέρας βίας. Κάτι ακόμη το οποίο είναι, είναι σημαντική πτυχή για την διατήρηση των αποθεμάτων είναι απόφαση διακοπής ε, των, ε, της αλίας ε, στο, στην ιστορική, στο ιστορικό ανώτατο όριο ή στο τρέχον επίπεδο, το οποίο είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή, 28 σκάφη δηλαδή, παραγαδιάρικα ισπανικά. Και μία ακόμη σημαντική πτυχή είναι το πολυμερές κομμάτι. Προβλέπεται ότι η συμφωνία δεν θα παραμείνει κλειστή, γιατί διέπεται από τα διεθνή ε, πρότυπα όλα τα αποθέματα δηλαδή ε, σε ιστορικά μέγιστα όρια ε, πρέπει να είναι ε, η διαχείρισή τους να γίνεται από κοινού, να γίνεται διεθνώς ειδικά όταν μιλάμε για την ανοιχτή θάλασσα και πρέπει να παραμένει ανοιχτά και σε άλλα κράτη όπως για παράδειγμα κράτη της Ασίας κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και σημαντική, σημαντικό αίτημα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα τέλος ε, να τονίσω ότι προβλέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας η δυνατότητα απόσυρσης, κοινής απόσυρσης ε, των εκκρεμών υποθέσεων και από τα δύο μέρη, των εκκρεμών υποθέσεων στο Διεθνές Δικαστήριο ε, για το Δίκαιο της Θάλασσας και στον ΠΟΕ, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί δύο υποθέσεις έχουν ανασταλεί από το 2000 ένα και κάθε χρόνο πρέπει να στέλνουμε επιστολές και στους δύο οργανισμούς και να εξηγούμε ότι θέλουμε να παρατείνουμε την αναστολή αυτή και η, η κατάσταση αυτή έχει συνεχίσει, συνεχίζει εδώ και πολύ καιρό και πιστεύουμε ότι είναι επιβλαβής και για τις σχέσεις μας ε, με την ε, χιλή γενικότερα, αλλά και την, ε, και βλάπτει και τη συνεργασία μας στην αλλιευτική με τη χιλή. Σε γενικό πολιτικό επίπεδο η συνεργασία με τη Χιλή είναι πολύ καλή και μόνο αυτό το πρόβλημα υπήρχε, το πρόβλημα με τον Ξηφία που ουσιαστικά είχε προκαλέσει ένταση στις ε, σχέσεις μας. Υπό τις διατάξεις αυτές ε, για την απόσυρση, ήδη από το Δεκέμβριο καταφέραμε να αποσύρουμε την ε, υπόθεση που εκκρεμεί στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας και ελπίζουμε να ε, αποσυρθεί και η υπόθεση ενώπιον του ΠΟΕ. Θα ήθελα επίση να πω ότι παρά το γεγονό ότι η υπόθεση θα αποσυρθεί, η υπόθεση που, έχει, που εκκρεμεί στον ΠΟΕ ε, θα αποσυρθεί, η υπόθεση για το TVR ε, θα παραμείνει εκκρεμή, γιατί υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με την εφαρμογή της συμφωνίας. Θα μπορούσαμε όμως, αν δεν, γίνει, αν δεν υπάρξει εφαρμογή, να ε, υποβάλουμε εκ νέου την υπόθεση στον ΠΟΕ, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, αν δεν θέλει να πάρει το λόγο κάποιος άλλος βουλευτής. Δεν ε, άκουσα να λέτε ότι όλα αυτά έγιναν το 1999 από μία ανακοίνωση που έγινε από την Διεθνή Ένωση των Ψαράδων με ε, ε, ε, παραγάδι, την Ανάπα. Ήταν σκάφη τα οποία μέχρι τότε αλίευαν χωρίς κανένα πρόβλημα αλλά προσέκρουσαν στην αντίσταση των χιλιανών αρχών όσον αφορά τη χρήση των λιμένων τους. Αυτό αντιβαίνει σε, όλα στα, σε όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και η Χιλή, ε, ενώ γνώριζε όλα αυτά, δεν ε, τηρούσε αυτούς τους κανόνες για εμπορικούς ε, λόγους και αυτός είναι ο λόγος για τους οποίους η ΑΝΑΠΑ προσέφυγε στον ΠΟΕ γιατί ήταν, αυτό ήταν ένα φραγμό στο εμπόριο. Εσείς είπατε ότι κατανοείτε ότι οι σχέσεις με τη Χιλή είναι καλές. Εκτός από αυτό το θέμα της αλίας του Ξηφία. Όχι, οι σχέσεις ήταν, δεν ήταν καλές γιατί δεν είναι καθόλου ευέλικτη χιλή σε θέματα αλίας. Όχι μόνο στο θέμα του Ξηφία, αλλά γέννη σε αληφτικά ζητήματα. Εγώ θα ήθελα επίσης να πω ότι οι διαβουλεύσεις που κάνετε σε σχέση με αυτό το μνημόνιο το 2009 ο κλάδος έκανε μια σειρά παρατηρήσεων σε σχέση με τους περιορισμούς που θέτει το μνημόνιο όσον αφορά την πρόσβαση στους λιμένες. Και εσείς βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ε, ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μονομερής ε, απόφαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά μια ελάχιστη πρόσβαση στους λιμένες της Χιλής. Και θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Ο τομέας... Εγώ δεν συμφωνώ να θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι, μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό εκ μέρους τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρόκειται για μια μονομερή απόφαση χωρίς ε, κανένα νόημα και θεωρώ ότι είναι καλύτερο να παραμείνει η προσφυγή στον ΠΟΕ και να ληφθεί μια απόφαση κατά πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αποδεκτό ή όχι γιατί σε άλλες περιπτώσεις ε, λέγεται στο μνημόνιο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις ε, ε, λιμένες, η Αρίκα, η φαγκάστα και η Πούντα Ρένες για την εκφόρτωση του ξηφία κλπ. Αλλά πρόκειται για παραγάδια άρικα σκάφη. Και μόνο το 50% αυτών των σκαφών ελιεύουν τον ξηφία είναι, νομίζω ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Ε, και σε σχέση με τον ανεφοδιασμό των ε, σκαφών, εκεί αναφέρονται επίσης κάποιοι περιορισμοί. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις από κάθε άποψη είναι εξαιρετικά περιοριστικές και από την έννοια αυτή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι σύμφωνη με αυτό το μνημόνιο, δεν συμφωνώ να αποσυρθεί, να η προσφυγή στο ΜΠΟΕ και από την άποψή μου είναι προτιμητέο να περιμένουμε την απόφαση του ΠΟΕ πριν αποδεχθούμε αυτό το μνημόνιο που όπως σας είπα όσον αφορά τη χρήση των λιμένων παραμένει προβληματικό. όσον αφορά τους ε, κανόνες που ισχύουν για τα σκάφη της ε, Χιλής που έρχονται στους δικούς μας λιμένες. Τα ύδατα αυτά ρυθμίζονται από την ε, ΣΕΑΤ που είναι διεθνής οργανισμός. Η Χιλή δεν είναι συμβαλόμενο μέρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος στον οργανισμό αυτό, αλλά όχι Χιλή. Και όσον αφορά το μνημόνιο του 2001, όπου η Χιλή έλεγε ότι θα ήθελε να υπάρξει ένας άλλος περιφερειακός οργανισμός της Αλίας όπου θα συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι πάντοτε βάζει εμπόδια στις συναντήσεις που γίνονται για την δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει να συγκληθούν, να, η, να γίνουν συνδυάσεις και οι διαβουλεύσεις για τη δημιουργία αυτού του νέου οργανισμού, η Χιλή προσπάθησε να το εμποδίσει. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να αποδεχτώ αυτό το μνημόνιο και θα ήθελα να αποσυρθεί έως ότου οι προϋποθέσεις ε, θεωρούνται αποδεκτές. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Εγώ λέω όλα όσα σκέφτομαι κύριε Καντέκ. Το θέμα αυτό το γνωρίζω καλά εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό έχω την ε, πολυτέλεια να πω αυτό το οποίο πιστεύω. Εγώ έχω ιστορική μνήμη. Είμαι σαν τα μαμούθ. Είμαι εδώ από την ε, εποχή της προϊστορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλετε μπορείτε να παρέμβετε κύριε Καντέκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε να είστε σκιώδη συγγήτρα σε αυτή την έκθεση, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά και γιατί αγαπάτε πολύ και τη Χιλή. Το κατάλαβα. Εγώ αγαπάω πολύ τη Χιλή, ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ με τα μαθήματα Ελίας που επιθυμούν να μας δώσουν οι Χιλιανοί. Θέλει κανείς άλλος να παρέμβει. Όχι, μιλάω σοβαρά, είναι ένα σημαντικό θέμα. είναι σημαντικό και σχετίζεται με τον ΠΟΕ. Η κυρία εκπρόσωπος της Επιτροπής επιθυμεί να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον Ισπανικό αλλιευτικό κλάδο, τους εκπροσώπης του Ήταν δύσκολα τα πράγματα στο φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου συζητήσαμε τη Σύμφωνη γιατί ήταν μια διαδικασία που έλαβε χώρα σε προεκλογική περίοδο στην ε, Χιλή και συνεπώς ε, ο αλληλευτικός ε, κλάδος επηρέασε τα πράγματα. Ήταν πολύ εχθρικό ως προς την συμφωνία αυτή. Δεν πρόκειται λοιπόν να επανέλθω σε αυτό. Αλλά όσον αφορά σε αυτό που αναφέρατε ότι 50% των αλλιευμάτων είναι, ξυφή, είναι ξυφίας και τα υπόλοιπα είναι άλλα ήδη μπορεί. Αλλά η εντολή που είχαμε εμείς και τα αιτήματα των κρατών μελών ήταν να διαπραγματευτούμε συμφωνία για τον ξυφία. Και αυτό κάναμε. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση Ήτλος, είπατε κι εσείς ότι για μας είναι Φραγμό στο εμπόριο, δεν είναι θέμα διατήρησης αποθεμάτων και το γεγονός ε, ότι υπήρχε μία υπόθεση στο πλαίσιο του Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας ήταν ε, μία υπόθεση που είχε να κάνει με την έλλειψη συνεργασίας ε, που ισχυρίζεται ότι υπήρχε, ισχυρίζεται η Χιλή ότι υπήρχε όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων του Ξηφία. Για μας όμως ήταν ένα ζήτημα φραγμός εμπορίου και γι' αυτό ο ΠΟΕ είναι αυτός που θα έπρεπε να επιληφθεί. Ευχαριστώ. Μου διευκρινίσατε και κάτι που δεν ήξερα. Ήταν και προεκλογική χρονιά στη Χιλή. Κατάλαβα γιατί έγινε η διαπραγμάτευση. Ε, αυτό μου είχε διαφύγει. Καλά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, διότι ο κύριος Γκάλαχερ δεν είναι εδώ. Θα του δώσουμε τις παρατηρήσεις που έγιναν εδώ. Στη συνέχεια έχουμε το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Κανόνες εισαγωγής από τη Γρυλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιθονόζων, δαθαλασσίων γαστερόποδων και υποπροϊόντων τους. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δόθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση συντονιστών και επειδή κανένας δεν το ήθελε, καμία πολιτική ομάδα, το πήρε η πρόεδρος. Η πρόεδρος θα κάνει το θέμα αυτό ως πρόεδρος και όχι ως κυρία Φράγα. Η Κομισιόν έχει το λόγο λοιπόν για να μας παρουσιάσει την πρόταση. Έχουμε εδώ Το λόγο ε, θα δώσουμε πρώτα στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο κυρίους που είναι εδώ θα παρέμβει. Ε, εσείς αποφασίστε ποιος θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ και μετά θα το δώσω στη Γενική Διεύθυνση Μάρε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει αυτή την πρόταση κατόπιν ετήσεως των κυβερνήσεων της Δανίας και της Ιρλανδίας. Το σκεπτικό είναι η Γρυλανδία να μπορεί να συμμετέχει στην ενιαία αγορά για την ε, παραγωγή ε, στην Ιγλανδία. Δεν μιλάμε μόνο για α, ψάρια, αλλά και για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ε, καθώς και παραπροϊόντα τα οποία προκύπτουν από αλληλεία και αλευτικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν ε, καλύπτονται και τα δίθυρα μαλάκια και τα υπόλοιπα είδη που αναφέρονται στην πρόταση. Αυτό γίνεται επί τη βάση μιας δέσμευσης αφενός ότι η ιδανική κυβέρνηση θα εποπτεύει και θα ελέγχει τις προ... υποχρεώσεις ε, που επιβάλλονται στη Γρυλανδία και οι υποχρεώσεις είναι ότι η Γρυλανδία θα μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα αλληλευτικά προϊόντα αυτά ή την παραγωγή τους. Αυτό, όπως βλέπετε στην πρόταση, περιλαμβάνει όχι μόνο τα πρότυπα παραγωγής ε, για την διατροφική ασφάλεια, αλλά και θέματα ε, υγείας των ζώων, όταν μιλάμε για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να ε, τηρηθούν τα πρότυπα παραγωγής για υποπροϊόντα όπως τα ηφθιέλεια ε, καθώς επίσης και τους κανόνες εισαγωγές να υπάρχει ένας, ένα σημείο ελέγχου των συνόρων στη Γρυλανδία και να συμμετέχουν και στα συστήματα ε, επικοινωνίας μέσω υπολογιστών τα οποία έχουν ε, συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία των ζώων και τον έλεγχο των ε, ζωικών προϊόντων και την εμπορία του στην ενιαία αγορά. Αυτή λοιπόν είναι η υποχρέωση την οποία έχει η Γρυλανδία και η ιδανική κυβέρνηση ε, και οι ιδανικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις ε, εφαρμογής και επιβολής ε, αυτής της υποχρέωσης. Πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το διάβασα, δεν διαπιστώνω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάπου στην πρόταση αυτή. Επομένως θα ετοιμάσουμε τη σχετική γνωμοδότηση και αν υπάρχει κάποια αμφιβολία θα διαβουλευτούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο και με αυτό να περάσουμε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 Bueno, pues a ver qué hacemos. La presentación. ¿Eh? Ahí viene κυρία Πατράου. Eh, Ωραία λοιπόν, η εισηγήτρια είναι εδώ, η κυρία Πατράου. Στο σημείο 10 λοιπόν τη ημερήσια διάταξη έχουμε τη Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ίσων ε, του Σολομόντο. Η εισηγήτρια, όπω σα είπαν η κυρία Πατράου, να δώσω το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει την παρουσίαση για τη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Φοντάνα εξ ονόματος Επιτροπής νομίζω. Δεν είναι καλής από την Επιτροπή εδώ. Τώρα μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα έρθει ο κ. Φοντάνα. Κυρία Πατράου, εσείς θέλετε να πείτε κάτι ή δεν θέλετε. Τι να σας πω, υποδιάλυση τελούμε. Εγώ έχω ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αφού δεν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορώ να τι σε εσά. Α, ήρθε ο κύριο Φοντάνα. Καλωσορίσατε, κύριε Φοντάνα. Άντε, καθίστε. Καλώς ορίσατε λοιπόν κύριε Φοντάνα. Μην ανησυχείτε, είμαστε μαθημένοι εδώ. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν είναι λίγο διαλυμένη. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία αλευτική σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και νήσων του Σολομόντος. Θα σας δώσω το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίαση πριν ακούσουμε τους ευρωβουλευτές και κατόπιν θα σας διατυπώσουμε κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προφανώς έφτασα την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να σας κάνω μερικά εισαγωγικά σχόλια σε σχέση με την συμφωνία αυτή και να απαντήσω βεβαίως ε, σε τυχόν ερωτήσεις. Ε, συνεπώς, ε, η Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νήσων Σολομόντος είναι τμήμα των συμφωνιών που έχουμε στον Ειρηνικό. Στο Δυτικό Ειρηνικό συγκεκριμένα έχουμε πολύ πλούσια αποθέματα τόνου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική τα αλληλεύματα τόνου είναι το ίμιση σχεδόν των αλλιευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αλλία μας. Όπως γνωρίζετε έχουμε τρεις συμφωνίες, ε, έχουμε και με το Κυριμπάτι και με την ε, μακρονησία ε, συμφωνίες εκτός από ε, τις συμφωνίες με τα νησιά Σολομόντος ε, μονογραφήθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 βάσει εντολής βέβαια από πλευράς ε, Συμβουλίου δύο πτυχέ, όπως όλες και οι συμφωνίες, μία πτυχή που αφορά την πρόσβαση και μία, αφορά, μία πτυχή που έχει να κάνει με την υποστήριξη της αλλιευτικής, ε, των, της των νήσων Σολομόντος. Εκτός λοιπόν από την πρόσβαση στα δικά μας σκάφη, πρέπει να ενισχύσουμε και τη συνεργασία μας με, τα, ε, με τις νήσους Σολομόντος και να ενθαρρύνουμε αηφόρο αλλιευτική πολιτική και υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων από ε, τις νήσους Σολομόντος. Τρία χρόνια θα διαρκέσει η συμφωνία και δίνει τη δυνατότητα, αλλιευτική, την αλλιευτική δυνατότητα για ε, ε, ισπανικά και γαλλικά, όχι όμως παραγαδιάρικα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποια ευελιξία, αν χρειαστεί, να εισαχθούν. Τώρα, όσον αφορά το τονάζ, 4.000 τόνοι, δηλαδή μείωση, γιατί ήταν 6.000 ε, στην προηγούμενη συμφωνία. «400.000 ευρώ είναι το κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν όντως ε, ε, διατεθεί οι πόροι αυτοί για την στήριξη της αλληλευτικής αυτής συμφωνίας και για τις δύο πτυχές που ανέφερα προηγουμένως. Κάτι ακόμη το οποίο έχει να κάνει συγκεκριμένα με τη συμφωνία αυτή είναι ότι έχουμε λοιπόν προσπαθήσει να εξυγχρονίσουμε κάποιες από τις διατάξεις της ε, σύμφωνα με βάσει των ε, ε, υπολείπων αλλιευτικών συμπράξεων. Θα δείτε δηλαδή μια ρήτρα που υπάρχει, μας δίνει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε δηλαδή κάποια τμήματα της συμφωνίας. Υπάρχει δυνατότητα αναστολής εφαρμογής της συμφωνίας ε, υπό συγκεκριμένε συνθήκες, αν για παράδειγμα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την εφαρμογή από την άλλη πλευρά της αλλιευτικής πολιτικής, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε σε αναστολή. Αν δεν υπάρχει συμφωνία κατανόηση μεταξύ ημών και των νήσων Τσολομόντος και επίση ε, έχουμε ενισχύσει τις διατάξεις όσον αφορά τα επιστημονικά στοιχεία και τις ε, επιστημονικές συμβουλές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ήδη για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη πίεση δεν είναι αντικείμενο υπεραλίευσης. Υπάρχει και μία ρήτρα ακόμη που είναι ε, κοινωνική, κοινωνικά ουσιαστικά, κοινωνική ρήτρα για ε, τις νήσους 25% των ναυτικών προέρχονται από τις ε, χώρες ΑΚΕ. Μετά τη μονογράφηση λοιπόν, Εμεί προετοιμάζουμε την απόφαση για την έναρξη ισχύω τη συμφωνία. Καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο λόγω τη έναρξη ισχύω της συνθήκης Λισαβόνα. Είναι η πρώτη ε, συμφωνία ελευτικής σύμπραξη ε, που ευθυγραμμίζεται με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπέβαλε στο Συμβούλιο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι επικείμενη η συμφωνία από πλευρά Συμβουλίου, και κατά τις επόμενες ε, ημέρες θα υποβληθεί και στο Κοινοβούλιο. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. Sí, Ευχαριστώ πολύ. Οι συμφωνίες αυτές, όπως ε, υπόθηκε, είναι πολύ σημαντικές για τον ε, τομέα της αλίας στην ε, κοινότητα, γιατί παρέχουν νέες ελευτικές ευκαιρίες και ακούσαμε κάποιους αριθμούς που πραγματικά αντανακλούν την κλίμακα, εκφράζουν την κλίμακα αυτών των ευκαιριών και δείχνουν πόσο σημαντικές είναι. Αλλά επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα ψάρια που μπορούν να ληφθούν και εμπέπτουν σε αυτή τη συμφωνία. Συμφωνώ, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αξιολογήσει αυτές τις συμφωνίες ελέγχθη ότι αυτή είναι η πρώτη αλληλευτική συμφωνία η οποία θα εμπίπτει στην συνθήκη της Λισαβόνας και διαπέτει από τους δικούς της ε, κανόνες. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι υπάρχει λόγος να, υπάρξει, να γίνει αναθεώρηση της ε, συμφωνίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και να υπάρξει συμφωνία κατά γράμμα. Οι επενδύσεις που συνεπάγεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοιου είδους συμφωνία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε στην ε, κοινή γνώμη υπό την έννοια των ενδιαφερόμενων πολιτών της εν λόγω χώρας, στην περίπτωση αυτή των ίσων του Σολομόντος. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να διευκρινιστούν εδώ και τα οποία μου ήρθαν στο νου καθώς διάβασα το κείμενο και τα οποία αναφέρθηκαν και στην παρουσίαση προηγουμένως. Ακούσαμε για μία μείωση από 6.000-4.000 τόνους. Στην ε, προηγούμενη συμφωνία δεν είχαμε απλώς πρόσβαση για τα λευτικά σκάφη του τόνου, αλλά για τα παραγαδιάρικα γενικώ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει, δεν ισχύει και την ε, νέα συμφωνία. Παρ' όλα αυτά ε, το κόστος είναι το ίδιο 400.000 ευρώ. Συνεπώς λοιπόν εγώ οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία αυτή μας δίνει λιγότερα. Έχουμε μία μείωση από 600.000-400.000 ε, τόνους, ο αποκλεισμός ε, των παραγαδιάρικων και παρόλα αυτά πληρώνουμε το ίδιο κόστος. Σε, σε σχέση με αυτό έχω να κάνω και δύο άλλα σχόλια φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν τα παραγαδιάρικα σκάφη εφόσον ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο οι ελείς των παραγαδιάρικων δηλαδή ενδιαφέρονται για την πρόσβαση των νήσων Σολομώντα ε, βεβαίως με το ίδιο κόστος δεν ξέρω, θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος στην περίπτωση αυτή. Νομίζω ότι είναι σαφές. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Φαίνεται ότι η συμφωνία που ισχύει μέχρι το 2009, που ισχύει μέχρι το 2009, δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή προς εμάς όσον αφορά τη σχέση αποτελεσματικότητας και κόστους. Εάν τα σκάφη του αλεύσης του τόνου ε, τους χορηγήθηκε άδεια μόνο σε 7 σκάφη και αν δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα ύδατα αυτών των λιμένων, αν δούμε τον όγκο της αλληλευτικής ικανότητας, νομίζω ότι δεν ε, ε, πληρούνται εξαντλείται αυτή η αληφτική ικανότητα. Ένα άλλο θέμα αφορά την συνεδρία της κοινή Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί αλλά δεν έλαβε χώρα. Τώρα θα ήθελα να μου... και θα ήθελα να μου πείτε γιατί, να μου αναφέρετε τους λόγους. Θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν εκεί. Και τέλος, ορισμός των ε, προϋποθέσεων ε, συνεργασίας με τις νήσους αυτές. 30% δίδονται στην ε, υποστήριξη της ατομικής πολιτικής στην νήσο. Αλλά δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για το πώς θα εφαρμοστούν αυτά, σε τι ακριβώς αναφέρονται αυτά τα 30%. Και έχω την άποψη ότι είναι ζωτική σημασία για μας να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των συμφωνιών και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πλήρης και αυστηρή εφαρμογή των συμφωνιών. Εάν το κάνουμε, για να το κάνουμε θα πρέπει να ξέρουμε ε, τι περιλαμβάνει ακριβώς το 30% αφορά την τομεακή πολιτική, την αλευτική πολιτική στα νησιά, δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. κυρία Eh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την κυρία Πατράου για τα ε, ενδιαφέροντα ερωτήματα που έθεσε. Έχω ένα ερώτημα σε σχέση με τους αλληλευτικούς πόρους ε, τόνου. Είπατε ότι περάσαμε από του 6.000 στου 4.000. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, Είναι επειδή τα αποθέματα του τόνου βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση. Η κατάσταση είναι σταθερή, δεν υπάρχει καμία υπεραλίευση. Γιατί αυτή είναι η αρχή στην οποία βασίζονται οι διάφορες ε, ε συμφωνίες. Δηλαδή, να μην ε, ε, διατίθενται πόροι που δεν μπορούν ε, οι αρχές της χώρας με τις οποίες κάνουμε τη συμφωνία να εκμεταλλευτούν. Όσον αφορά τώρα την υποστήριξη της τοπικής αλίας, θα ήθελα να μάθω αν κάνατε αξιολόγηση του τοπικού αυτού αλλιευτικού κλάδου. Και αν κάνατε αξιολόγηση, σε τι ακριβώς ε, θα χρησιμεύσει η υποστήριξη αυτή στην τοπική αλία και όπως είπε και η κυρία Πατράο, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο αυτή η μεικτή επιτροπή δεν συνεδρίασε. Θα ήθελα να μάθω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλές σχέσεις ε, με τις νήσεις Σολομόντος. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια, γιατί και εγώ ε, στον καιρό μου είχα ασχοληθεί με αυτή τη συμφωνία Λίας. Θα ήθελα να ρωτήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί λέτε ότι πρέπει να ε, τα προσαρμόσετε στη ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2004, διότι ήδη είχαμε συμφωνία εταιρική σχέσης γιατί πρέπει να τα προσαρμόσουμε στα συμπεράσματα του 2004. Εγώ πριν από τρία χρόνια απασχολήθηκα με αυτή τη συμφωνία, ήταν συμφωνία εταιρική σχέση. Τι ακριβώ ε, θα προσαρμόσουμε, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, θεωρώ θετικό σε σχέση με τις επικρίσεις που είχε κάνει στην προηγούμενη συμφωνία με τα νησιά του Σολομόντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γεγονός ότι έχουν εισηχθεί κάποιες από τις παρατηρήσεις μας στη νέα συμφωνία. Και θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικός ο διαχωρισμός του κόστους ε, στο κόστος για τις αλευτικές δυνατότητες, δηλαδή αποσημείωση για αυτό το οποίο καταβάλλεται, το οποίο αυτή τη στιγμή χωρίζεται. Έχουμε 240.000 ευρώ για τις αλευτικές δυνατότητες και τα υπόλοιπα δίνονται ως ε, συνδρομή για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Γίνεται λοιπόν διαχωρισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων σε σχέση με τα υπόλοιπα και αυτά ήταν ένα από τα αιτήματα τα οποία είχαμε διατυπώσει. Γι' αυτό λοιπόν με χαροποιεί το γεγονό ότι έχει συμπεριληφθεί. Κάποιες άλλες επικρίσεις που είχαμε ήταν το θέμα των ε, ναυτικών οι οποίοι έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τα θυναλιευτικά τα οποία έχουν συγκεκριμένες συμφωνίες και ε, δεσμεύονται από συγκεκριμένες συμφωνίες διότι ο τόνος είναι μεταναστευτικό είδος και έχουν συγκεκριμένες άδειες και ο καθένας πρέπει να λιεύει βάσει των αδειών που διαθέτει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έλυσε με κάποιους κανόνες οι οποίοι λένε ότι καθορίζεται ένα ποσοστό χωρών και επομένως ρυθμίζεται το πρόβλημα το οποίο είχαμε στο παρελθόν. Βέβαια, πρέπει να συνεχίσω να επικρίνω δύο πτυχέ οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και εδώ διαφωνούμε. Το πρώτο είναι το θέμα των ε, συμβαλωμένων. Ξέρω ότι σε αυτή την περίπτωση οι συμβαλόμενοι είναι για να έχουμε κάποιους εδώ αλλά ούτε ο ε, τομέας τους θέλει, ούτε κάποιος άλλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν ε, ε τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν όταν δεν τους θέλει κανείς. Δεύτερον, το θέμα των παρατηρητών. Δεν είναι κανεί κατά των παρατηρητών. Αυτό το λέω εκ των προτέρων. Αλλά στην προηγούμενη συμφωνία για να έχουμε παρατηρητέ έπρεπε να καταβάλλονται 400 ευρώ ένα σκάφο. Και τώρα αυτό το ποσό αυξήθηκε και πήγε στα 1500 ευρώ. Υπερτριπλασιάστηκε. Το κόστο ζωή ε, τη νήσου του το Σολομώντα δεν φαντάζομαι να τριπλασιάστηκε. Γιατί λοιπόν γίνεται τόσο μεγάλη αύξηση και μάλιστα αυτό καταβάλλεται όταν γίνεται η αίτηση. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς πρόβλημα έχουν οι χώρες, μας, οι χώρες αυτές με τους ε, εφοπλιστές μας. Αυτό το ποσό πρέπει να το καταβάλουν ε, οι νήσοι του Σολομόντα και από εκεί και πέρα ο εφοπλιστής πρέπει να καταβάλει τα έξοδα διατροφής κλπ το κάθε σκάφος θα πρέπει να το καταβάλει ε, αυτό το ποσό ενώ όλοι δεν έχουν παρατηρητές επί του σκάφους. Δεν το καταλαβαίνω ακόμα αυτό το θέμα των παρατηρητών. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να ε, παίρνουμε χρήματα επιπλέον από τους εφοπλιστές χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα μου εξηγήσετε για ποιο λόγο έγινε αυτή η αύξηση από τα 400 στα 1500. Εάν μου απαντήσετε με κάποιο εύλογο εγώ επιχείρημα δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά πρέπει να μου το εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτή η άξιση. Ε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ο, η κυρία Ανδρέας Μπαρέα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα ζητήσει και πριν το λόγο. Δεν με είδατε μάλλον. Τρεις ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη έχει να κάνει με τη μείωση στους ε, τόνους. Ε, ως επιχείρημα προβάλλεται η επιστημονική αξιολόγηση και λέτε ότι αυτό γίνεται βάση επιστημονικών αξιολογήσεων. Ισχύει αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Στην προηγούμενη συμφωνία η Ένωση των Επιχειρήσεων λειτουργεί, ε, δεν λειτουργεί... Ε, προβλέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η ένωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Και τρίτον, το θέμα της παράνομης αλίας. Πώς ε, διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες και πώς διεξάγεται τους συγκεκριμένους ελέγχους. Νομίζω ότι αυτά είναι συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα μας δώσουν μια πλήρη εικόνα. Νομίζω ότι ε, είναι καλά τα στοιχεία που έχουμε στο έγγραφο που παρουσιάζεται, ε, αλλά αυτά τα στοιχεία θα συμπληρώσουν ευνοϊκά την εικόνα που έχουμε. Ο κύριος Φοντάνα. Thank you. So, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Θα αρχίσω με την ερώτηση που έχει να κάνει με την αξία, με το κόστος της ε, συμφωνίας αυτής και νομίζω ότι υπήρξαν και πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Στις διαπραγματεύσεις ε, η μείωση του τονάζ αναφορά ε, έλαβε υπόψη ε, πολλά στοιχεία. Δεν είναι μόνο το ένα στοιχείο, ένα στοιχείο που καθόρισε ε, τον αριθμό αυτό. Μία από τις πτυχέ είναι η επιστημονική, τα επιστημονικά στοιχεία. Υπάρχουν ορισμένα είδη τόνου που υφίστανται πιέση και επομένως έπρεπε να μειωθεί βάσει των επιστημονικών δεδομένων η τόνη αλίευση. Κάτι ακόμα. Αυτό αντικατοπτρίζει τα αλλιεύματα από τον αλλιευτικό στόλο των προηγούμενων ετών. Κάθε φορά που κάνουμε διαπραγμάτευση πρέπει βεβαίως να αξιολογήσουμε τα αλλιεύματα και την ε, χρήση των ε, ε, αλλιευμάτων της περασμένης χρονιάς. Κάθε φορά που υπάρχει μείωση, ή μεταξύ του τονάζ και των αλλιευμάτων βάσει της συμφωνίας και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και γι' αυτό ακριβώς υπήρξε μείωση ε, των ε, τόνων. Όσον αφορά τώρα το κόστος, ο λόγος που έχουμε το ίδιο κόστος αλλά μικρότερο τον ζω, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ότι θέλαμε να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την υποστήριξη της τομεακής πολιτικής περισσότερο από τις προηγούμενε προηγούμενες ε, συμφωνίες σύμπραξη. Συνεπώ, Συνεπώς, αν θέλουμε λοιπόν να αντισταθμίσουμε τη μείωση αλλίευση τόνων με τη χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, της υποστήριξης της ε, ε τομεακής πολιτικής στις είναι ένας τρόπος ε, να ε, γίνει αυτό. Από πλευράς λοιπόν εμπορικής, ε, για να το πω έτσι, υπάρχει βέβαια μία μείωση της, ε, του κόστους, αλλά από ως αναπτυξιακής, δηλαδή από πλευράς αηφόρου αλλιευτική πολιτικής, υπάρχει μεγαλύτερη αξία για τις νήσους Σολομόντος και αυτό εντάσσεται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τις, την αηφόρο αλλία στις τρίτες χώρες. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο στοιχεία τα οποία Κάπω αντισταθμίζουν το ένα το άλλο. Όσον αφορά στους παρατηρητές, αυτό ήταν κατόπιν αιτήματο των νήσων Σολομόντο. Γνωρίζετε ότι σε γενικέ γραμμές τα προγράμματα παρατηρητών ε, την χάνουν χρηματοδότησης. Δεν νομίζω ότι αυτό δηλαδή αντανακλά κάποια αύξηση του ε, κόστους ε, ζωής ε, στις νήσους Σολομόντος. Απλώς προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη περισσότερο το κόστος των προγραμμάτων παρατήρησης που είναι σημαντικότερο, είναι μεγαλύτερο στον Ειρηνικό ωκεανό. Στο πλαίσιο, με των κατευθυντηρίων γραμμών, βάσει των οποίων ότι, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πλήρω αυτό το κόστο. Αυτό ήταν ένα αίτημα των νήσων Σολομόντος. Όσον αφορά την παράνομη αλία, πιστεύουμε ότι αυτή η αύξηση της ενίσχυσης στην τομεακή πολιτική στη χώρα θα τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση των προηγούμενων συμφωνιών, Υπήρξε ένα ερώτημα κατά πόσο αξιολογήσαμε τις την προηγούμενη συμφωνία. Βεβαίω το κάναμε και θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έγιναν διαπραγματεύσει που βασίστηκαν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση που έγινε από πλευρά ε, ε, Επιτροπή και υποβάλαμε και στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα αυτή. Έχουμε και το κείμενο, αν θέλετε να δείτε τι λεπτομέρειε αξιολόγηση προηγούμενη συμφωνία. Όσον αφορά τη μεικτή επιτροπή, γιατί υπήρξε ένα ερώτημα για ποιο λόγο δεν συνήλθε προηγουμένω. Ο βασικό λόγο είναι όπως γνωρίζετε, αυτές οι χώρες έχουν τη δυσκολία πρόσβασης. Δεν μπορούσαμε πριν από την ε, εκπνοή της ε, συμφωνίας ε, να πάμε. Όμως, στις διαπραγματεύσεις αξιολογήσαμε από κοινού με τις νήσου Σολομόντος την προηγούμενη συμφωνία. Το συζητήσαμε μαζί τους και αυτό και αυτό ελήφθη υπόψη στην σύναψη της συμφωνίας. Τώρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πώς θα καταβληθεί αυτό το ποσό, το 50% υπέρ της τομεακής πολιτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή συγκριθεί η συμφωνία από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο τότε θα γίνουν συζητήσεις ε, με τις ε, νήσους Σολομόντος ε, για να συμφωνήσουμε επί συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν ως τμήμα της τομεακής πολιτικής. Αυτό θα συζητηθεί στη Μικτή Επιτροπή με τη συμμετοχή των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου ως παρατηρητή. Θα υπάρξει λοιπόν ένας οδικός χάρτης για να το πω έτσι. Τι θα κάνουμε λοιπόν με τους πόρους αυτούς για την ανάπτυξη της τομεακής πολιτικής στο μέλλον. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με την συνάδελφο που αναφέρθηκε στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. Η έναρξη ισχύω της θα μας βοηθήσει να δούμε τις λεπτομέρειες της ενίσχυσης της τομεακής πολιτικής και όσον αφορά την τοπική αλληλεία, μάλλον δεν εξήγησα καλά, δεν μιλούσα για την τοπική αλληλεία, Μιλούσα για τους τοπικούς αλληλείς. 25% του, ε, ε, των ναυτικών ε, στα ε, πρέπει να προέρχονται από χώρες ΑΚΕ. Με προτίμηση αλληλείς των νήσων Σολομώντας. Δεν μιλάω λοιπόν για τοπικές επιχειρήσεις, μιλάω για τους, για τους αλληλείς. Και αυτό θα το λάβουμε υπόψη όταν θα χορηγούμε τις άδειες και θα το δούμε αυτό στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής. Το τελευταίο σχόλιο που είχε να κάνει με τα παραγαδιάρικα, ο λόγος για τον οποίο δεν διαπραγματευθήκαμε αλληλευτική δυνατότητα για τα παραγαδιάρικα είναι ότι στα προηγούμενα, τα τέσσερα χρόνια πριν από την διαπραγμάτευση ε, υπήρχε μηδενική χρήση των αδειών για τα παραγαδιάρικα και συνεπώς δεν θεωρούσαμε ότι δικαιολογεί το να συμπεριλάβουμε άδειε ε, στην ε, Συμφωνία σύμπραξη, Αν όμω υπάρξει ανάπτυξη ε, του ε, στην ε, περιοχή θα μπορούσαμε να το θέσουμε στα, στις νήσους Σολομόντος και να δούμε κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν άδειε και για τα παραγαδιάρικα. Αλλά εφόσον δεν, υπήρχαν χρησιμοποιηθεί, δεν είχαν χρησιμοποιηθεί άδειε στο παρελθόν δεν βλέπω το λόγο να γίνει διαπραγμάτευση για τα σκάφη αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα πρέπει να πω ότι συνεχίζω να έχω αμφιβολίες τρία σημεία όσον αφορά τα παραχαδιάρικα. Γνώριζα ότι το ποσοστό ήταν μηδέν στο παρελθόν αλλά το ερώτημά μου ήταν το εξή. Εάν αναπτυχθεί ο τομέα και αν υπάρξει ενδιαφέρον, κατά πόσο θα συμπεριληφθεί στο κόστος των 400 ευρώ η χρήση των γαδιάρικων. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, άκουσα τις εξηγήσεις που δόθηκαν ότι υπό τη νέα συμφωνία υπάρχει μία μείωση σε εμπορικό επίπεδο, αλλά λέχθη ότι υπάρχει μία αύξηση πόρους με όρους ανάπτυξης. Μου φαίνεται δύσκολο να καταλάβω εδώ τα επιχειρήματα. Έναν παρέχεται δύο επίπεδο χρηματοδότησης και τελικά μειώνεται η ελίευση. στις ευρωπαϊκές χώρες θα λέγαμε ότι πληρώνουμε τους ανθρώπους για να μην ψαρεύουν. Και αυτό είναι κάπως δύσκολο να το καταλάβουμε. Έπειτα η κοινή επιτροπή. Είπατε ότι είναι δύσκολο για την επιτροπή να συνέλθει και αυτό θα γίνει μετά τη θέση ισχύ της συμφωνίας. Για να δούμε πώς θα ρυθμιστεί η μεκι υποστήριξη εάν αυτό πράγματι ισχύει, τότε ε, πώς θα ρυθμιστεί αυτή η τοπική υποστήριξη. Αυτό θα πρέπει να συνδυθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Νομίζω ότι είναι... Εγώ συνεχίζω να έχω προβλήματα σε αυτά τα τρία θέματα. Ίσως η Επιτροπή θέλει να επανέλθει. Έχετε το λόγο. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Όσον αφορά τα τελευταία ερωτήματα, Βεβαίως ε, υπάρχει υποθετική αύξηση, αν υπάρξει υποθετική αύξηση του, της αλίας με παραγαδιάρικα θα πρέπει να αναθεωρηθεί η συμφωνία. Αυτό προβλέπεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για εισαγωγή αυτού του μέτρου. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με τις ε, πραγματικές αλληλευτικέ δυνατότητες. Ίσως η προηγούμενη αλληλευτική συμφωνία δεν μας έδινε, ε, δεν ήταν ε, σωστή η σχέση κόστους και απόδοσης. Τώρα υπάρχει ομερότερο κόστος για την πρόσβαση, παρόλο που δεν το βλέπουμε σε αυτά τα 400 ευρώ. Παρόλο που δίδεται περισσότερα χρήματα για την τομεική υποστήριξη, πρόκειται από τον προπολογισμό για τις ενίσχυση Σολομόντος, ε, το κόστος πρόσβασης στην πραγματικότητα είναι χαμηλότερο. Και αυτό λέφτε υπόψη στην, ε, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χαμηλότερης χρησιμοποίησης τα προηγούμενα χρόνια. Ε, θα υπάρξει λοιπόν μια αύξηση χρηματοδότησης της νήσους του Σολομώντα για την αλληλευτική τους πολιτική. Εάν το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουμε την τομεακή αλία στις νήσους Σολομόντος, η απάντηση είναι ότι ναι μεν θα αλεύουν τα ίδια ψάρια ή ελπίζουμε περισσότερο, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα να δίδονται περισσότερα κονδύλια για τη χάραξη της δικής τους πολιτικής, γιατί είναι τμήμα της δικής μας ε, προσπάθειας να υποστηρίξουμε μια βιώσιμη αλία. Ούτε Και νομίζω ότι μετά την απόφαση συμβολή αυτό θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται μόνο για μια εμπορική συμφωνία. Τέλος, για την ε, Κοινή Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι ναι, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε ε, να προτείνουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε τη συνήθεια του Σολομόντος πριν τεθεί σε συμφωνία. Άρα, επισήμως, οι στόχοι που πρόκειται να εγκριθούν σε σχέση με το μεκή υποστήριξη των νήσων του Σολομόντος, αυτό θα γίνει μέσω της μικτής επιτροπής, γιατί οι στόχοι συμφωνούνται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις νήσους. Δεν είναι δυνατόν πριν από τη σύγκληση αυτής της επιτροπής και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε αυτό να γίνει ε, σύντομα αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φοντάνα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Όχι, τότε έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη. Κυρία Λόβιν έχει το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαντήσατε στο ερώτημά μου για τη μείωση τη ποσόστοση στη συμφωνία που βασιζόταν σε επιστημονικά δεδομένα. Τώρα λέτε ότι πριν αλλιεύαμε την ίδια ποσόστοση αλλά πληρώναμε περισσότερο που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, χρησι... δεν ε, αξιοποίησε πλήρως αυτά για τα οποία είχε πληρώσει και τώρα έχουμε μειώσει την ποσόσταση επειδή υπάρχουν λιγότερα ψάρια στον ωκεανό αλλά λέτε ότι εξακολουθούμε να πληρώνουμε ε, όσο πριν. Άρα δεν καταλαβαίνω ποια είναι η μείωση. Κάνουμε υπεραλίευση αυτή τη στιγμή, γιατί αν μειώνονται τα αποθέματα και έχουμε το, την ίδιο αριθμό ποσοστώσεων με το παρελθόν, σημαίνει ότι κάνουμε υπεραλίευση τώρα. Πρέπει κάπως να μου το εξηγήσετε αυτό. Και κάτι ακόμη, όταν είπα τοπική ντόπια λύση ε, δεν ξέρω, μήπως ε, παρεξηγήθηκα, γιατί αναφέρθηκα στην υποστήριξη των εθνικών αλλιευτικών πολιτικών που θα έπρεπε βεβαίως να προωθεί τους ντόπιου αλλοίς κατά τη γνώμη μου. Αλλά βέβαια, αν υπήρξε αξιολόγηση, δεν ήταν μόνο αυτό το ερώτημά μου αν υπήρξε αξιολόγηση, ήταν, το ερώτημά μου ήταν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ικανοποιημένη με την αξιολόγηση αυτή και, και μιλάω για την προώθηση των ντόπιων αλλιέων στο πλαίσιο της προώθησης εθνικής αλλιευτικής πολιτικής. Ε, uh, Ωραία. Ζητώ συγγνώμη αν δημιούργησα σύγχυση με την αναφορά στο τονάζ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπεραλίευση στη συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι πριν υπήρχε δυνατότητα υπεραλίευση, διότι το συνολικό τονάζ αναφοράς ήταν υψηλότερο και αυτό χρειάστηκε να το μειώσουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχει υπεραλίευση. Τώρα, η διαφορά μεταξύ των πραγματικών αλευμάτων και του τονάζ υπάρχει, αλλά έχουμε μειώσει το τονάζ ώστε να μην υπάρχει κανένα ενδεχόμενο υπεραλίευσης. Αν το είχαμε αυτήσει στους 6.000 τόνους, και ο Ευρωπαϊκό Στόλο είχε εξαντλήσει αυτού του 6.000 ε, τόνου του τονάζ αναφορά, τότε θα είχαμε υπεραλίευση. Νομίζω ότι αυτό μα βοηθά να παρακολουθούμε την υπεραλίευση και μα επιτρέπει να βρισκόμαστε και εντό των ορίων που, των αλευμάτων που μπορούμε να αλλιεύσουμε. Τώρα, με το θέμα των ε, ναυτικών, ε, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια, θα πρέπει να το επανεξετάσω και να σας ενημερώσω. Μία μικρή διευκρίνηση λίγο αργότερα θα σας δώσω. Ε, θα αποφασίσει ο πρόεδρος βέβαια, αν μου επιτρέπει να το κάνω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, την εξαντλήσαμε την ε, πρωινή μερίσια διάταξη. Ε, λύεται η συνεδρίαση, αλλά σας υπενθυμίζω ότι τρει η ώρα έχουμε και κλεισμένο το θερόν ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις ε, τρει μέχρι τις τέσσερι και μισή και ξέρετε ότι αυτό αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Ευρωβουλευτές και τους Συμβούλους των Πολιτικών Ομάδων και τη Γραμματεία της Επιτροπής Αλίας. Όλοι οι άλλοι δεν επιτρέπεται να παρέμβουν. Ε, συνεχίζουμε στις 3.